Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μερικά προβλήματα στην ημερήσια διάταξη. για λόγους που υπέκφευγαν, διέφευγαν το ελέγχο μας, ε, συνθμήθηκε η απογευματινή ημερήσια διάταξη και ο εισηγητής ο κύριος Κάρθη που έχει το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη με τη γνωμοδότηση δηλαδή που αφορά το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη Μία και Μία Υγεία και την προσπάθεια καταπολέμησης της ε, μικρο... μικροβιακής αντοχής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ επιλαμβάνεται και μάλιστα είχαμε και τον Ιούλιο συζήτηση σχετική με τον Αρμόδιο Επίτροπο. Και τελικά αναβάλλεται στο σημείο για τις 21-22 Φεβρουαρίου. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη που έμεινε πολύ κουτσουρεμένη με ένα μόνο σημείο. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μετάδοση της συνεδρίασης απευθείας στο διαδίκτυο και διερμηνεί από και προς 20 γλώσσες με εξαίρεση τα τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και γοεδελικά. Σημείο 3, όπως είπαμε, αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 21ης 22ης Φεβρουαρίου. Περνάμε λοιπόν στο μοναδικό σημείο που μας έμεινε, το σημείο 4, την εφαρμογή του κανονισμού για το πρόγραμμα φυτοπροστασίας. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Γιάρ που συντάσσει γνωμοδότηση, γιατί δεν είμαστε η αρμόδια καθήλια επιτροπή, απλώς γνωμοδοτική επιτροπή. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι η αρμόδια κατουσία για το θέμα αυτό και εμείς θα επιδώσουμε τη γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Και μάλιστα όταν έγινε η διαπραγμάτευση για τον κανονισμό και κατόπιν ε, εγκρίθηκε το 2006, τότε η Επιτροπή μας έλαβε το καθεστώς της Συνδεδεμένης Επιτροπής και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι βασικοί χρήστες ε, των ε, προϊόντων φυτοπροστασίας και εξαρτημένη από τη διαθεσιμότητα ε, επαρκών, κατάλληλων και σε προσιτές τιμές προϊόντων φυτοπροστασίας. Οι κύριοι δικαιούχοι και εξαρτημένοι από αυτό είναι οι γεωργοί. Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος ζητήθηκε από το Γραφείο Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την ομάδα της μεταγενέστερης αξιολόγησης ε, έκθεση εμπειρογνωμοσύνης. Αυτή η έκθεση ανατέθηκε σε έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα που εκλήθη να αξιολογήσει το σημερινό επίπεδο εφαρμογής του κανονισμού και επικεντρώνεται κυρίως στην ικανότητα των κρατών μελών να δίνουν αξιόπιστες άδειες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μια χαρτογράφηση των πρακτικών της επιστημονικής αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν στα κράτη-μέλη. Ο εισηγητής της γνωμοδότησής μας είναι ο κύριος Γιάρ, που απουσιάζει όμως σήμερα και εκπροσωπείται από τον κύριο Ντες. Ο κύριος Αλφρεντές, λοιπόν, εκ μέρους του ηγετή γνωμοδότηση του κυρίου Γιάρ, θα μα παρουσιάσει την έκθεσή του για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι ο Πατεριάρη είναι πάντα πάνω στην Επιτροπή μας, όμως δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μου έδωσε το σημείωμά του να σας το διαβάσω και να τον εκπροσωπήσω και μας λέει ότι όπως ορίζει και το χρονοδιάγραμμα 26 Ιανουαρίου έχουμε την προθεσμία και κατάθεση των τροπολογιών ψηφοφορία στην Επιτροπή για τις 23-24 Απριλίου ψηφοφορία στην Ολομέλεια από ό,τι προβλέπεται το 2018, μέσα στο 2018 και όπως είπε και ο πρόεδρος αρμόδια κατ' ουσίαν είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος με τον κύριο Μποκ από τους σοσιαλιστές δημοκράτες. Τώρα στα γενικά σχόλια, ο Πέτερ Γιάρ ε, εκφράζει τη λύπη του ότι στη δημόσια συζήτηση δεν γίνεται λόγος επαρκώς για τους ε, κινδύνους από τα φωτοπροστατευτικά προϊόντα διατυπώνονται μόνο, για τα φωτοπροστατευτικά προϊόντα γίνονται, διατυπώνονται μόνο κατηγορίες και πολλές φορές παραγνωρίζει κοινή γνώμη την πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν ταυτοπροστατευτικά προϊόντα για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των τροφίμων και να μην καταστρέφεται η εσόδια. Οι γεωργοί στο μεγαλύτερό του ποσοστό υποστηρίζουν αυστηρέ νομοθετικέ διατάξει και για την πιστοποίηση και για τη χρήση, έτσι ώστε αρνητικέ συνέπειε για το περιβάλλον, τον, τη δημόσια υγεία και τα ζώα να αποφεύγονται. Η δουλειά των γεωργών δεν θα πρέπει να ε, κινδυνεύει από φοβικές αντιδράσεις ε, αλλά να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Η εναρμόνιση των συστημάτων πιστοποίησης των αυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει επιτέλους να προχωρήσει. Χρειάζονται κριτήρια για ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει ούτε αυτό, ούτε, διαθε... ούτε εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους γεωργούς. Δεν πρέπει να υπάρχουν ειδικέ λύσεις σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται στην Ευρώπη ένα ενιαίο σύστημα διατάξεων ώστε να αποφεύγονται και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Και εδώ μου επιτρέπετε μια προσωπική παρατήρηση μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε διατυπώσει το αίτημα στην Ευρώπη να ε, ρυθμιστεί το ζήτημα των προστατευτικών προϊόντων με ένα κανονισμό ε, με πιο αυστηρές διατάξεις σε σχέση με αυτά που μέχρι τώρα ήταν δυνατά σε εθνικό επίπεδο. σε ορισμένα κράτη δηλαδή υπήρχαν αυστηρέ διατάξει, δεν έχω ακριβώ τα νούμερα και τα ονόματα, αλλά αυτό είχε σαν συνέπεια στη Γερμανία περίπου 8% των αυτοπροστατευτικών ουσιών να απαγορεύονται, ενώ ε, μέχρι και 24% των ίδιων των ουσιών ε, θα μπορούσαν να απαγορευτούν σε άλλα κράτη, γιατί ήταν διαφορετικά τα συστήματα πιστοποίηση. Η πιστοποίηση αδειοδότηση θα πρέπει βεβαίω να βελτιώνει και την διαθεσιμότητα και την ε, ποιότητα, την προστασία δηλαδή των διαφόρων ειδών, φυτικών ειδών, ώστε να περιοριστεί και ο όγκος των εισαγωμένων φυτικών προϊόντων. Αντίστοιχα αιτήματα μας διατυπώνουν και οι γεωργοί της Βαβαρίας. καθώς και το αίτημα να ενισχυθεί το ζήτημα της έρευνας στα προστατευτικά προϊόντα, γιατί οι παραγωγοί κατασκευαστές των προστατευτικών προϊόντων δεν είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν πολλά εκατομμύρια για την έρευνα. Ε, πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί ποιότητα, καλά γεωργικά προϊόντα, με εγγυημένη ποιότητα. Η τήρηση των νομοθετικών διατάξεων με μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ε, νοσοκόνων παραγόντων είναι απαραίτητη σε ενιαίο επίπεδο. Στόχος του κανονισμού θα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων, σε σχέση με την χρήση των φωτοπροστατευτικών και στην γνωμοδότηση διατυπώνεται το ερώτημα αν επιτυγχάνεται με τις λύσεις που έχουν προταθεί ε, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα της γνωμοδότησης είναι ότι δεν εξασφαλίζεται. Περνούν ακόμη και 120 μέρες μέχρι να εξασφαλιστεί η άδεια για ένα ε, προϊόν για το οποίο έχει ζητηθεί αδειοδότηση σε ορισμένες περιοχές, ενώ σε άλλες ε, χώρες είναι πολύ πιο σύντομα τα υπόλοιπες ε, τομέ οι προθεσμίες καθώς είναι χωρισμένη σε ζώνε Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες. Τα κράτη-μέλη δυστυχώ δεν εφαρμόζουν όπω πρέπει τον κανονισμό. Η κατανομή εργασία μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να προχωρήσει κατά τρόπο οργανωμένο, μεθοδικό. Έχουμε τέσσερις ε, κρατικές αρχές και δύο διαφορετικά ε, υπουργεία αρμόδια για το θέμα αυτό μόνο στη Γερμανία. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και βέβαια η πληθώρα οργανισμών και φορέων που είναι αρμόδιοι οδηγούν σε αδιαφάνεια στην αγορά. Αυτά λοιπόν εκ μέρους του Πέτερ Γιάρ ο οποίος ε, μας δηλώνει πως είναι τεθμένος να εξετάσει τις ε, τροπολογίες και να δεχθεί ε, τόσ, εκείνες οι οποίες αποβαίνουν σε όφελος τόσο των γεωργών όσο και των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ξεκινούμε από τους και ηγητές. Κυρία Μακεντάερ, από το ECR που επήγεται να λάβει πρώτα το λόγο γιατί έχει και άλλη συνεδρία στην οποία θα πρέπει να μεταβεί. Παρακαλώ έχετε το λόγο κυρία Μακεντάιρ. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω τώρα γιατί πρέπει αργότερα να πάω στην Επιτροπή Απασχόληση για να παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου. Καταρχήν αναγνωρίζω ότι ο κανονισμό 1107 ε, είναι αρμοδιότητα καθήλη τη επιτροπή περιβάλλοντο, Εξού και η, σημασία, η μεγάλη σημασία αυτή τη γνωμοδότησης Επιτροπής Γεωργίας γιατί εδώ και εμείς μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τις απόψεις των γεωργών και να δώσουμε φωνή στους γεωργούς ε, τονίζοντας τις ανάγκες τους. Γι' αυτό και είναι σημαντικό η Επιτροπή ΕΜΒΗ να λάβει υπόψη τη δική μας γνωμοδότηση για τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Ευχαριστώ θερμά τον Πίτερ για το έργο του. Ε, αντιλαμβάνομαι πλήρως ε, τα όρια στον αριθμό των λέξεων που ισχύουν για τις γνωμοδοτήσεις και παρά τα μικρά περιθώρια. Ήταν πολύ αξιόλογο το πόνημα του κυρίου γιάρκη. και ελπίζω με τις τροπολογίες μου να το εμπλουτίσουμε περαιτέρω. Είναι ανησυχητικό που από την έγκριση του κανονισμού 1107 καταφέραμε μόνο να δώσουμε άδεια για πέντε νέες δραστικές ουσίε. Και είναι πολύ ανησυχητικό που συρρυκνώνεται τόσο πολύ η εργαλειοθήκη των γεωργών. Ουσιαστικά στερούνται αποτελεσματικών και χαμηλοκίνδυνων προϊόντων και έτσι εξαρτώνται από μικρό ρυθμό προϊόντων φυτοπροστασίας με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη γλυφοσάτη. Θα ήθελα να απευθύνω μια ιδιαίτερη έκκληση για τις περιορισμένες χρήσεις και τις ειδικές καλλιέργειες. Ακριβώς ε, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής μου, τα απορροκυπευτικά είναι πολύ σημαντικός κλάδος της γεωργίας. Και ουσιαστικά μιλούμε για καλλιέργειες ειδικέ που απαιτούν ε, ίσονες χρήσεις. Δεν δώσαμε όμως αρκετά κίνητρα και ενάυσματα στον κλάδο ε, για να λάβει άδεια έγκρισης ε, για τέτοια προϊόντα και το Ταμείο των ε, Περιορισμένων Χρήσεων δυστυχώς δεν ανταπεξήλθε στην αποστολή του. Και θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες ως προς το θέμα αυτό για να επικεντρωθούμε σε αυτές τις ισονές ε, χρήσεις και τις ειδικέ καλλιέργειες. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιο είναι το μέλλον της αγροτεχνολογίας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε νομοθεσία και έγκριση των προϊόντων φυτοπροστασίας που να είναι κατάλληλοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Γιατί έχουμε ε, drones και ρομπότ ή κάποια, κάποιες συσκευέ ρομποτικής που περιορίζουν τη χρήση της φυτοπροστασίας. Μπορούμε λοιπόν να συντεριάξουμε τον τρόπο χρήσης των προϊόντων φυτοπροστασίας με τις ε, ποσότητες και τις διαδικασίες για την πιστοποίησή τους. Επίσης θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την παράγραφο 3 που τονίζει τη μεγάλη σημασία μιας ε, επιστημονικής προσέγγισης της πολιτικής μας. Είναι σημαντικό λοιπόν η πολιτική μας να δράζεται σε επιστημονικά πορίσματα, να εξετάσουμε μελέτες ανάλυσης κινδύνου και μελέτες επιπτώσεων και αντικτύπου και να εδράζουμε τις αποφάσεις μας σε επιστημονικά πορίσματα και αποδείξεις και όχι σε κάποιες ε, ακραίες απόψεις που μερικές φορές ε, ε, υιοθετούνται ή εκφράζονται. Ευχαριστώ θερμά τον Πίτερ Γιάρ και θα έχετε να την στην υποστήριξή μου στην διεκπαιρέωση της γνωμοδότησής του. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον Πίτερ Γιάρ για την έκθεσή του. Και επίσης και στο συνάδελφο από την παρουσίαση ήταν λίγο δύσκολο γιατί ε, υπήρξε, κάποια, είχαν, υπήρξε μια σύγχυση ανάμεξη κάποιων στοιχείων τα οποία ήταν στην αρχική, είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική γνωμοδότηση. Ε, η Επιτροπή αυτή και η γνωμοδότηση ασχολείται με την γεωργία και όπως αναφέρει ο τίτλος και με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δηλαδή υπερβαίνει τα όρια των ε, επιχειρήσεων ε, παραγωγής ε, προϊόντων και θεωρώ ότι αυτό το έχει συμπεριλάβει ο Πέτερ Γιάρ, δηλαδή το ζήτημα της ανάπτυξης της υπαίθρου και της δυνατότητας για τους γεωργούς να ζήσουν και να εργάζονται στο χώρο της υπαίθρου. Όταν μιλάμε για την ε, φυτοπροστασία, η εμβέλεια της ε, φυτοπροστασίας την οποία χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Γεωργία αλλά και σε σχέση με την ε, χρήση στο δημόσιο χώρο καθώς και την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε τέτοιου είδου ε, δραστικές ουσίες ε, στο πλαίσιο των ιδιωτικών ε, νοικοκυριών. Αυτή είναι η άλλη πτυχή. Όλοι αυτοί οι παράγοντε θα καθορίσουν το, την εμβέλεια τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η φυτοπροστασία λοιπόν από τη μία πλευρά σημαίνει ότι καταστρέφεται η ζωή. Και θα ήθελα να το δω ε, στο πλαίσιο του συνόλου, της συνολικής ε, γεωργίας την οποία έχουμε. Γιατί δεν, ε, η μη συνετή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι δυνατόν να παρεμποδίσει και να βλάψει, να καταστρέψει το υπέδαφος, την ατμόσφαιρα κλπ. Ε, και βεβαίως υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι κάνουν βιολογική γεωργία αλλά τελικά ε, μολύνονται οι δικές βιολογικές καλλιέργειες από τους ε, συμβατικούς καλλιεργητές οι οποίοι χρησιμοποιούν βλαβερά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επίσης το θέμα της ποιότητας των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει εδώ να το εξετάσουμε. Όταν μιλάμε για την επιστημονική πρόσβαση, βεβαίω υποστηρίζω πλήρω αυτή τη δυνατότητα. Αλλά θα ήθελα να σα υπενθυμίσω μια συζήτηση που έχει γίνει. Δηλαδή, το ζήτημα είναι ε, ποια θα πρέπει να είναι η ποιότητα τη επιστημονική τεκμηρίωση και των επιστημονικών μελετών, ούτω ώστε να έχουμε έναν επαρκή βαθμό διαφάνεια κατά την διενέργεια αυτών των ε, μελετών και τη ε, συλλογή επιστημονικών στοιχείων. Ένα άλλο θέμα είναι η σωρευτική επίδραση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο κίνδυνος ε, δεν προέρχεται μόνο από το σύνολο των επιμέρους ε, ζυζανιοκτώνων, αλλά ε, προέρχεται από την σωρευτική δράση μιας συστηματικής χρήσης τέτοιων ουσιών. Και από την έννοια αυτή θα επαβάλουμε κάποιες εμπληρωματικές τροπολογίες στο σχέδιο αυτής της νομοδότησης και θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίω τον Πέτερ Γιάρ για την πολύ καλή συνεργασία που υπήρξε επικοδομητική ήδη από πέρσι. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Κάντεμαχ, η κυρία Σκοτ Κάτω έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και λυπούμε που έφυγε η κυρία Μάκεντάρ, γιατί θέλω να αναφερθώ σε κάποια από τις δικές παρατηρήσεις είπε καταρχάς ότι ρόλο μα είναι να υποστηρίξουμε του γεωργού και μια ειδική κατηγορία γεωργικής παραγωγή. Ναι, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι και του καταναλωτέ, όπω και τους παραγωγούς τροφίμων πρέπει να υποστηρίζουμε. Αυτό είναι καθήκον μας, όπως άλλωστε είναι καθήκον μας να υποστηρίζουμε κάθε τύπο παραγωγού και όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν την υψηλή τεχνολογία. Επίση θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση την οποία βλέπει η κυρία Μάκιντάρ να πρόκειται για ένα νέο πόλεμο των κόσμων δεν υπάρχει ένας νέος πόλεμος των κόσμων, κάτι τέτοιο φαίνεται να βλέπει. Η διαδικασία διοδότης λοιπόν των ζυζανοκτώνων στη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόσφορη. Θα πρέπει να γύρουμε διάφορα σημεία που μας ανησυχούν μέσα από την έκθεση, από την γνωμοδότηση και χαίρο που έχει την έκθεση καθήλυνη η ΕΝΒΗ, αφορά και τη δική μας δουλειά βέβαια εδώ στην ε, Επιτροπή Γεωργίας οι επικαλύψεις, οι μη δημοσιευμένες εκθέσεις και μελέτες ε, μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα και ως καθηγήτρια έχοντας εργαστεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ε, βεβαίως ξέρω ότι χρειάζεται και πρέπει να υποστηρίξουμε αμερόληπτες εκθέσεις και μελέτες και όχι κάτι που έχει χρηματοδοτήσει ο ίδιος ο κλάδος με βάση τα συμφέροντά του και το ίδιο ισχύει και για την αδειοδότηση. Το είδαμε άλλωστε και στην ε, υπόθεση της ε, γλυφωσάτης όπου δεν δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή τεράστιος όγκος στοιχείων ε, πάνω στα οποία είχαν στηριχθεί οι ε, μελέτες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια Επιτροπή εξεταστική για τη γλυφωσάτη να αναπτύσσεται και ε, ταυτόχρονα τη διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατόν κατά την αδειοδότηση να στηριζόμαστε σε αντικειμενικά στοιχεία, σε μερόληπτες μελέτες, με συνέπειες σοβαρές και για τη βιοπικιλότητα και για το περιβάλλον, όπως και για τη δημόσια υγεία μες των τροφών που καταναλώνουμε. Πρέπει λοιπόν να είναι φυσικά προϊόντα τα ζωνιοκτώνα να μην στηρίζονται σε, σε αμφίβολη σημασία, αξίας μάλλον ε, χημικά και αυτά εφόσον είναι έτσι δεν θα πρέπει να περνούν από την ε, δύσκολη αυτή διαδικασία της αδειοδότησης για να μπορούσαν να παραμένουν και βιώσιμα. Φυσικά συνθετικά χημικά ή ε, γενικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της αδειοδότησης. Ε, πρέπει να εξετάζονται συνέπειες σε ε, είδη του ζωικού βασιλείου, τα οποία δεν στοχεύει καταρχήν το Ζανιοκτών όπως τα νοικοτονοειδή, από ό,τι ξέρουμε βλάπτουν ε, τον πληθυσμό της, ε, των μελισσών. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέπεται και επιπλέον, αν πρόκειται για διαδότη σε περίπτωση εξαιρετική ή έκτακτη ανάγκη, αυτή πρέπει να είναι όντω έκτακτη και εξαιρετική και όχι να γίνεται γενικευμένη χρήση για λόγου άλλου. Κατά τα άλλα, θα υποστηρίξουμε τη γνωμοδότηση με τι τρομοδότησει. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φλάναγκαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την γνωμοδότηση και τη συζήτηση. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Σκοτ το Ποιον υπηρετεί η Επιτροπή μας, η Επιτροπή μας υπηρετεί όποιον καταναλώνει τροφή ουσιαστικά δηλαδή όλους τους πολίτες. Ε, μπορούμε να έχουμε υπόψη ακόμη και εκείνο το καταναλωτή ο οποίος μπορεί να μην έχει γεωργική παραγωγή, να μην ζει σε αγρόκτημα, αλλά να ζει στην πόλη και να καταναλώνει τα γεωργικά προϊόντα. Βεβαίω και πρέπει να υποστηρίζουμε τους γεωργούς και να τους βοηθούμε ε, στον βιοπορισμό του, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να Εξασφαλίστε το συμφέρον το γενικό, το δημόσιο συμφέρον και όχι μόνο το καθενός το ειδικό, ιδιαίτερο συμφέρον. Δεν μπορούμε να λέμε είμαστε Γεωργική Επιτροπή και άρα υποστηρίζουμε τους γεωργούς μόνο. Όχι, δεν υποστηρίζουμε μόνο τους γεωργούς, αλλά γενικότερα και την ανάπτυξη της υπαίθρου και όλους τους καταναλωτές και δεν μπορούμε να έχουμε μια μονοδιάστατη προσέγγιση. Ε, κάτι ακόμη που βρίσκω ενδιαφέρον στη γνωμοδότηση είναι μια προσέγγιση η οποία είναι πολύ ουδέτερη ως προς ε, ε, τη σήμανση των προϊόντων και σε αυτό δυσκολεύομαι πάρα πολύ γιατί όταν είχαμε πει για τα σιγαρέτα ότι ε, θα αφήσουμε την σήμανση στους παραγωγούς το σχόλιο που είχε ακουστεί ναι, ναι, για φανταστείτε όμως ένας κατασκευαστή σιγαρέτων να βάλει σήμα πάνω στο πακέτο καπνίζεται όσο είστε γκέι γιατί κάνει καλό στο παιδί σα, Αυτό έχει δείξει το παράλογο τη κατάσταση. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε σε θέση ω Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν πρόκειται να χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα, φερειπίν την εσωπονία, εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει χρήματα με τι επενδύσει, τη, θα πρέπει να έχει και εκείνη ένα μάτι, μια εξέταση, να μπορεί να εξετάζει δηλαδή πού πάει αυτή η επένδυση στην πατρίδα μου, την ιδιαίτερη, γίνονται επενδύσει, οι οποίε αν αποτέλεσμα έχουν έχουν τη ρήπανση των ποταμών και την καταστροφή του φυσικού τοπίου. Ε, καταστρέφουμε τα, χρήματα, ε, ποτάμια μας με χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ας γνωρίζει λοιπόν η δεξιά την πράτη αριστερά και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένες και οι δύο με το ένα και ενιαίο μυαλό και αυτό σημαίνει α μην δίνουμε τα πάντα στι ε, επιχειρήσει. ας κοιτάξουμε και τον απλό πολίτη. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Μάλιστα. Ακούσαμε τους και ηγητές. Περνάμε στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Χόισλινγκ. <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ παρά να πω ότι συμφωνώ με την προλαλήσασα. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε εδώ μια επιτροπή η οποία εκπροσωπεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των καλλιεργητών γιατί έτσι δεν θα μας πάρει κανείς σοβαρά. Όσον αφορά τη η γνωμοδότηση του κυρίου Γιάρ, ε, εδώ δεν άκουσα ούτε λέξη για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην φυτοπροστασία. Ε, εάν κατάλαβα καλά, ε, δεν θα πρέπει να μπερδέψουμε την προστασία του περιβάλλοντος και τη φυτοπροστασία. Αλλά ελπίζω να μην κατάλαβα καλά, γιατί δεν ήταν τώρα ένας συζητητής να γνωρεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια Υπάρχουν επιστημονικές ε, έρευνες οι οποίες ε, δείχνουν για παράδειγμα ε, πως τα αποδημητικά πουλιά χάνουν το δρόμο τους λόγω αλλαγών στο περιβάλλον, στη φύση. Αλλά δεν μπορεί ο συγκτής να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. και ένα άλλο θέμα όσον αφορά την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Δεν υπάρχει η επιστήμη όπως δεν υπάρχουν η πολιτική, αλλά υπάρχει μια κάπως διαφοροποιημένη εικόνα. Δηλαδή από τη μία υπάρχουν πολλές πλευρές, δεν υπάρχει μία, μία και μοναδική επιστήμη, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, αποκλίνουσες επιστημονικές ε, απόψεις. Και υπάρχει το πρόβλημα ένας ολόκληρος επιστημονικός ε, κλάδος να έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και να χρηματοδοτείται, να πληρώνεται από εκείνους οι οποίοι επιθυμούν ε, τελικά να πάρουν την έγκριση για αυτές τις δραστικές ουσίες. Δεύτερο, δεύτερο σημείο. Ε, λέγεται ότι δεν θα εγκρίνονται νέες δραστικές ουσίες. Ναι, ε, αυτό το λένε και ενώσεις ε, γεωργών, ότι δεν, δεν, δεν υπάρχουν νέες θαυματουργές ε, ε ουσίες οι οποίες ε, μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά ως ζυζανιοκτώνα για την καλλιέργεια της κράμβης για παράδειγμα. Ε, η Γεωργία έχει σπαταλήσει όλα τα πυρομαχικά. Ωστόσο, στον κανονισμό αυτό αναφέρεται ότι οι καλλιεργητέ θα πρέπει να ψάξουν κάποιες εναλλακτικέ δυνατότητε πριν στραφούν στα ζυζανιοκτώνα. Και μεταξύ αυτών των εναλλακτικών ε, ε, δυνατοτήτων είναι η αμυψισπορά. Και και πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι της ε, αύξησης της ε, μικροβιακής ανθεκτικότητας. Και ε, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ ο εισηγητής βρίσκεται σε εντελώ λάθος τροχιά και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να παρέμβουμε διορθωτικά σε αυτή την έκθεση. Γιατί αν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά τους εαυτούς μας θα πρέπει να ασχοληθούμε τα προβλήματα που αφορούν την απώλεια της βιοπικιλότητας και την αύξηση, γιατί το βλέπουμε των ε, ζημιών για το περιβάλλον. Ε, και θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται ε, όσον αφορά την αρμόνιση της νομοθεσίας. Η νομοθεσία όσο έχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γι' αυτό θα υποβάλουμε και τις δικές μας τροπολογίες και μπορείτε να φανταστείτε ότι θα πάνε προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Αλλά ελπίζω τελικά να πετύχουμε ένα συμβιβασμό στον οποίο να μπουν και άλλα στοιχεία και όχι μόνο αυτή η πλευρά της κόπα κοτσέκα. Παρακαλώ να μην υπερβαίνετε το τρίλεπτο όσοι λαμβάνετε το λόγο. Κύριε Αγγιλέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ, για να προσθέσω και εγώ λίγα στοιχεία στην έκθεση πρωτοβουλίας και τη γνωμοδότηση του κυρίου Γιάρ, να πω ότι κάποιες προτάσεις του κυρίου Γιάρ είναι ενδιαφέρουσες, μερικές ε, θα τις συμπληρώσω με τις τροπολογίες μου. Ε, συνεχίζοντας αυτά που είπε ο κύριος Χόισλινγκ, θα ήθελα να πω ότι εδώ συνεχίζουμε την παραγωγή με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στις 25 χρόνια έχουμε καταργήσει 700 δραστικές ουσίες από τη χρήση. Μέσα σε 25 χρόνια απαγορεύσαμε 700 δραστικές ουσίες ουσιαστικά δεν μπορούμε πια να τι χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 700 δραστικές ουσίε. Και αυτό είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 700 δραστικές ουσίε ε, απαγορεύθηκαν. Και από τότε που τέθηκε ενισχύ ο κανονισμός έχουν δοθεί άδειε μόνο για 5 τέτοιε δραστικές ουσίε. Είναι προφανέ λοιπόν ότι έχουμε μια αισθητή μείωση σε ό,τι αφορά το ρυθμό των εγκρίσεων και τη χορήγηση αδειών για δραστικέ ουσίε. Και καλό θα ήταν να διαβρύνουμε κάπως τη γνωμοδότηση του κύριου Γιάρ, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Παρόλο που αναγνωρίζεται ε, αμοιβαία, υπάρχει η αναγνώριση της διαδικασίας αμοιβαία αναγνώριση, δεν χρησιμοποιείται αυτή η αμοιβαία αναγνώριση, γιατί υπάρχει δυσπιστία μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονό ότι κάποια χώρα στο σύστημά τη ε, επιτρέπει ε, τη χρήση μια δραστική ουσία δεν είναι αρκετό για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μια άλλη χώρα. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχει δυσπιστία και επιφυλακτικότητα μεταξύ των χωρών, οπότε δεν λειτουργεί αμοιβαία αναγνώριση. Πολύ καλό το μέτρο που λέει ο κ. Γιάρα, αλλά αναποτελεσματικό, μια και δεν εφαρμόζεται. Κάθε χώρα δεν εμπιστεύεται τις αξιολογήσει των άλλων χωρών και κρίνει σκόπιμο να κάνει και τη δική τη αξιολόγηση. Και αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα. Γι' αυτό είναι και τόσο περίπλοκη διαδικασία, γιατί δεν εφαρμόζεται η αμοιβαία αναγνώριση. Ίσως χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό γραφείο ε, γενικής καθολικής αναγνώρισης, γιατί σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου κυριαρχεί η δυσπιστία, η καχυποψία απέναντι στα συστήματα αξιολόγησης, ε, ακόμη και δυσπιστία απέναντι στις επιστημονικές αναλύσεις. Όντως, ε, ασκήθηκαν κριτικές ε, στα επιστημονικά πορίσματα και είναι πιθανό κάποιοι επιστήμονες να επηρεάζονται από τους χρηματοδότες τους. Αλλά εδώ έχουμε θεσμικά όργανα και σε εμά θα πρέπει να πριτανεύει η γνήσια επιστημονική ανάλυση. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι για να γίνει αποτελεσματική η αμοιβαία αναγνώριση, θα πρέπει να εφαρμόζεται. Και αν υπάρχει δυσπιστή και καχυποψία, α δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού τη αμοιβαία αναγνώριση για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Γιατί υπάρχει μια καθολική δυσπιστία που μα απαρεμποδίζει Είμαστε τόσο ε, απαιτητικοί απέναντι στους δικούς μας γεωργούς για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Αλλά δεν είμαστε αντίστοιχα απαιτητικοί από του ε, υπόλοιπου. Γιατί τέτοιε δραστικέ ουσίες που εμείς έχουμε απαγορεύσει, εφαρμο, ε, ε, εφαρμόζονται στα προϊόντα τρίτων χωρών και εμείς εισάγουμε προϊόντα με τέτοιες απαγορευμένες σε εμά ουσίες. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε το σύστημα της αναγνώρισης, να ισχύσει αμοιβαία αναγνώριση και να είμαστε εξίσου απαιτητικοί απέναντι και στις εισαγόμενα προϊόντα. Θα υποβάλλω και τροπολογία, γιατί δεν μπορούμε μόνο να απαγορεύουμε δραστικές ουσίες χωρίς να δίνουμε εναλλακτικέ λύσεις και έτσι να κόβουμε ε, τις ε, επιλογές των γεωργών. Ευχαριστώ. Ο Χαίτεμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ εκπροσωπώ τον, την σκιώδη συγκήτρια της ομάδας των φιλελευθέρων, την κυρία Μίλλορ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω εκ μέρους της ε, κυρίας Μίλλορ τον κύριο Γιάρ, ε, γιατί η το σχέδιο γνωμοδότησής του αποτελεί εξαιρετική βάση για τις μετέπειτα εργασίες μας. Ε, ε, επισημαίνει τις βασικές αδυναμίες του 1107 και την εφαρμογή και διαπιστώνει ότι λόγω έλλειψη εναρμόνιση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Υπάρχουν συστηματικέ καθυστερήσει στη διαδικασία έγκριση των δραστικών ουσιών με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένε χρήσει των έκτακτων πιστοποιήσεων και εγκρίσεων με αποτέλεσμα να στερούμε από του ε, γεωργού πολλά εργαλεία. Ο βασικό σκοπό του 1107 είναι να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων και να καταστήσει συμβατή τη γεωργία με το περιβάλλον. Επίση, η επιστημονική προσέγγιση για την αδειοδότηση των προϊόντων φυτοπροστασία έχει συγκεντρώσει επιθέσεις και κριτική τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε ένα πρόβλεπτο περιβάλλον για τους ε, παρασκευαστές. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια διορατική προσέγγιση με έμφαση στην καινοτομία της φυτοπροστασίας εν ώψη των τη μελλοντική μεταρρυθμίση του 1107 και για να βελτιώσουμε του στόχου και την υλοποίηση των στόχων του κανονισμού, θα πρέπει οι Γεωργοί να έχουν πρόσβαση σε, ένα, σε μια ευρεία εργαλειοθήκη δραστικών ουσιών, ώστε να μπορέσουν να, να ε, αντιμετωπίσουν του επιβλαβεί οργανισμού. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να μειώσουμε και τι δραστικέ ουσίε. Θα πρέπει να δώσουμε ενάβσματα και κίνητρα για την καινοτομία Γι' αυτό και θα καταθέσω σχετικέ τροπολογίε. Επίση, θα πρέπει να βρούμε και στον κανονισμό αυτό τρόπους για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη προ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίηση και Αδειοδότηση και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια των Τροφίμων. Την έφυσα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αντριέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο για, για την έκθεσή του. Δεν ακούγεται δυστυχώς πολύ καλά το μικρόφωνο του κυρία Αντρία, γιατί μιλάει μακριά από το αναμένο μικρόφωνο. Ε, εκπλήσωμαι πάντως που ο εισηγητής δεν λέει τίποτα για την παρούσα διαδικασία που χρησιμοποιείται ε, για την ε, προγενέστερη της άδεια ε, φάση. Γιατί είχαμε χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γλυφοσάτη γιατί έχουμε την κατάσταση του τότος κράτους, της Επιστημονικής Επιτροπής, της ανεξάρτητης μελέτης. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που είναι κάπως συγκεχημένα. Και έχουμε και την προσέγγιση της επιτροπολογίας, με την οποία πια είμαστε εξοικειωμένοι. Όλα αυτά θα πρέπει να ε, συμπεριληφθούν στην έκθεση και στην ανάλυση. Αναφέρθηκε, αναφέρθηκε ο νέος άνεμος που εισπνέει πια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της αδειοδότηση, αναγνωρίζονται σε αδυναμίες του κανονισμού 1107. Αλλά και ο κεντρικός κανονισμός 178 του 2002, που επίσης ε, περιέχει αδυναμίε. Την περασμένη εβδομάδα ε, ζητήσαμε μια καλύτερη ανάλυση για να διαλευκάνουμε τη διαδικασία θέση σε εμπορία των προϊόντων φυτοπροστασίας. Επίσης, είναι προφανές ότι θα πρέπει να μειώσουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων, ώστε να εγγυθούμε όλο και μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας και της υγείας και του περιβάλλοντος. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την ευθύνη που έχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, να εξασφαλίσουμε διαφάνεια σε όλες τις φάσεις εξέτασης ε, και εφαρμογή, ε, καθώ και να εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα των επιστημονικών εργασιών που αποτελούν τη βάση των πολιτικών μα αποφάσεων. Ευχαριστώ. κυρία Σάιρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω ευχαριστώ τον Πέτερ Γιάρ και όλου και όλε συντάκτες. Ε, συμφωνώ με τα σχόλια, με διάφορα από τα σχόλια που ακούστηκαν. Ε, είναι σημαντικά και ε, υπάρχει ένα ψήφισμα του 2017 όπου με τις τροπολογίες μας είχαμε ζητήσει να δοθεί έμφαση σε νέα προϊόντα, λιγότερο ρυπογόνα, ιδιαίτερα για, το, για τα ύδατα. Γι' αυτό με διαδικασία κατεπήγουσα. Μέχρι τώρα η κατεπήγουσα αυτή διαδικασία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Είναι πολύ σημαντικό όμως το θέμα αυτό για μας, καθώς πρόκειται για ζητήματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που βεβαίως είναι χρήσιμα για τους καλλιεργητές, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τηρηθεί αυτή η δέσμευση και η υπόσχεση. Δεν ε, μεριμνούμε μόνο για τους γεωργούς, μιλούμε για όλο το χώρο της φύσης και της γεωργίας και μέχρι και της μέλησης, αλλά και για όλους τους πολίτες που ζουν στις περιοχές αυτές της υπαίθρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ο κύριος Νταντάν τον συναρφό Γιάρ. Πολύ εύστοχα επεσήμανε κάποια από τα ζητήματα. Όπως πήγε η κυρία Αγγιλέρα, ωστόσο, θα ήθελα και εγώ να ξανακοιτάξουμε το ζήτημα της αμοιβαία αναγνώρισης και της ε, διάθεσης νέων αδειών ε, για ε, κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά. Βεβαίως είχαμε στηρίξει πολλές ελπίδες στο κείμενο αυτό που θα έπρεπε και τις διαδικασίε να επιταχύνει και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών και διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν επιτεύχθη. Πρόκειται για αποτυχία. Η αδειοδότηση για διάθεση στην αγορά θεωρείται από πολλούς πως έχει μπει στο σιρτάρι και δεν ξέρουμε πότε θα δοθεί. Ε, δεν έχει αποκατασταθεί εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών, γιατί όπως πολύ εύστοχα επισημάνθηκε νωρίτερα, ε, συνεχίζει ο καθένας ε, να κάνει τις δικές του μετρήσεις, αμφισβητώντας τις μετρήσεις του γειτονά του. Είναι απαραίτητο, πιστεύω, να έχουμε ένα νέο κείμενο, ένα κείμενο το οποίο θα δίδει την ευρωπαϊκή διάσταση στις ε, διαδικασίες αυτές και που θα καλύπτει και τις μαύρες τρύπες. Τι είναι οι, μικρές, οι μαύρες τρύπες, είναι η μικρή παραγωγή. Δηλαδή σήμερα έχουμε μια σειρά πολύ εξειδικευμένων ε, παραγωγών, παραγωγής, ε, που δεν προσφέρει προϊόντα γιατί είναι τέτοιες διαδικασίες που οι ε, επιχειρήσεις δεν καταθέτουν πια αιτήματα για αδειοδότηση. Και για πολλές από αυτές τις παραγωγές ε, έχουμε περιέλθει σε αδιέξοδο γιατί δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει έρευνα. Καθυστερούμε λοιπόν, καθυστερούμε σημαντικά και κινδυνεύουμε ακόμη κάποιες από τις παραγωγές αυτές να επαφεθούν σε άλλες περιοχές του κόσμου, οι οποίες για να είμαστε και ειλικρινεί, έχουν οπωσδήποτε ε, ελέγχους πολλά υπολοιπόμενους σε σχέση με αυτά που κάνουμε εμείς στην Ευρώπη και κινδυνεύουμε να αρχίσουμε να εισάγουμε τέτοια προϊόντα χωρίς έλεγχο, χωρίς να ε, υπάρχουν οι επαληθεύσεις ε, και με έναν ε, καταναλωτή ο οποίος θα τα αγοράζει ακόμα, ακόμα όχι μόνο αγνοώντας εάν είναι ασφαλή αλλά μόνο με την έννοια ότι βοηθάει χώρες πιο φτωχές ανά τον κόσμο. Είναι κάτι λέει, το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε. Ευχαριστώ. Thank uh, Θα ήθελα να θέσω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Το σύστημα ζωνικής ε, καταχώρησης το οποίο θέλουν να χρησιμοποιήσουν και κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή χώρα η οποία το εφαρμόζει θα πρέπει να τηρήσει την προθεσμία των 120 ημερών. Και το ερώτημά μου έχει ως εξή ε, ισχύει αυτό τώρα ε, ή ε, τελικά υπάρχουν καθυστερήσεις, εφαρμόζεται αυτή η προθεσμία, τηρείται. Όσον αφορά την αγώγηση της ασφάλειας των συνθετικών ζυζανιοκτώνων, είναι πολύ εύκολο να πει κανείς ε, ότι ε, δεν είναι ασφαλή γιατί ε, εάν βεβαίω χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες αυτών των επιβλεπών δραστικών ουσιών θα είναι μοιραίες συνέπειες. Και πάντοτε μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα θέματα αυτά είναι επικίνδυνα. Και αυτό βεβαίως υπονομεύει όλη τη διαδικασία. Διότι το θέμα είναι το ζήτημα του ρίσκου και όχι του κινδύνου και εξαρτάται από το ποια σκοπιά το εξετάζουμε. Ε, και υπάρχει ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού και εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτό οι οποίοι ε, χρησιμοποίησαν για πολλά χρόνια αυτές τις δραστικές ουσίες και το ποσοστό της έκθεσης ήταν χίλιες φορές παραπάνω από ό,τι για το συνήθι ε, καταναλωτή. Then of course If the European Union keeps banning these materials, Τέλος πάντων, εάν ε, συνεχίσουμε να απαγορεύουμε αυτές τις δραστικές ουσίες, τελικά θα αμοιαθεί η παραγωγή τροφίμων και θα εισάγονται, ε, οι δραστικές, θα εισάγονται τα τρόφιμα αυτά, τα οποία είναι μολυσμένα από δραστικές ουσίες, από άλλες χώρες του κόσμου. Άρα ε, ε, τα αποτελέσματα θα είναι απολύτω αρνητικά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια τροποποίηση σε αυτό το επιχείρημα γιατί είναι πιθανόν βεβαίως να έχουμε καλλιέργειες οι οποίες δεν χρειάζονται δραστικές ε, ουσίες. Ε, και επίση υπάρχει και το ζήτημα της απαγόρευσης των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών εκ μέρους αυτών που χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες η κυρία, η ομιλήτρια, μια προηγούμενη ομιλήτρια μίλησε για, την, ε, για τους ε, καλλιτές που κάνουν βιολογικές ε, καλλιέργειες και που δέχονται τις αρνητικές συνέπειες από τις συμβατικές καλλιέργειες. Ε, ε, οι, αυτοί που κάνουν βιολογικές ε, καλλιέργειες έχουν ε, μεγάλες ε, δυσκολίες να αντιμετωπίσουν ζυζάνια και ασθένειες στις βιολογικές καλλιέργειες και τελικά αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν, να εφαρμόσουν κάποιες μεθόδους που είναι επίσης μη θεμητές. Και βεβαίως ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φύση δεν είναι πάντοτε ούτε αγνή ούτε ε, ευεργετική. Οι φυσικές μέθοδοι καθηλέρειας. Η προηγούμενη ε, παρέμβαση θεωρώ ότι ήταν ανυπόφορη για μένα, αλλά δεν θα επισέλθω στα όσα υπόθηκαν. Θα αναφερθώ σε δύο σημεία τα οποία δεν αναφέρθηκαν. Το ένα είναι το ζήτημα της ευθύνης δεν υπάρχει ξεκάθαρη ευθύνη όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και πιστεύω ότι εάν θέλουμε μακροπρόθεσμα να έχουμε μια σωστή νομοθεσία θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ζήτημα της ευθύνης γιατί δεν είναι δυνατόν για να αυξηθεί η σοδιά να χρησιμοποιούνται κάποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ε, ε, και, αλλά παραμένει ασαφές θα γίνει όταν οι ουσίες αυτές καταλήξουν για παράδειγμα στον υδροφόρο ορίζοντα. Θα πρέπει λοιπόν το ζήτημα της ευθύνης να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησή μας, γιατί ε, πρόκειται για ουσίες που, των οποίων τις επιπτώσεις δεν μπορεί κανείς να τις οριοθετήσει ή των οποίων τις καταστροφικές συνέπειες δεν μπορεί να τις πληρώσει, να τις ε, διορθώσει. Δεν υπάρχει μια ανεξάρτητη έρευνα επιστημονική υπόθηκε. Εγώ θα έλεγα ότι οι οικολογικές οργανώσεις εδώ θα είχαν ε, αντιρρήσεις. Ε, οι μόνοι οι οποίοι είναι ύποπτοι τελικά είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες οι οποίοι χρηματοδοτούν ε, την έρευνα προκειμένου να στηρίξουν τις δικές τους θέσεις. Μια ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα είναι απολύτως αναγκαία και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει η σχετική επένδυση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. λέγεται ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες ε, βιολόγων οι οποίοι ε, ε, δεν και ε, ε, ασχολούνται με αυτά τα δηλητήρια τα οποία είναι πραγματικά δηλητήρια, δεν είναι απλώς ε, τοξικές ουσίες. Και μία λύση εδώ θα ήταν να υπάρχει μία φορολόγηση των ζυζανιοκτώνων. Είναι μία λύση που εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες. Ε, άλλους τους κάνει πραγματικά να τους σηκώνονται οι τρίχες. γιατί ίσως είναι επιζήμιες για ορισμένους ε, κλάδους, αλλά για τον καταναλωτή μια τέτοια φορολόγηση θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη. Ο Δενανό, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Πέτερ Γιάρ, γιατί πραγματικά οι προτάσεις του συνιστούν εξαιρετική βάση για τη συζήτηση. Θεωρώ ότι η μείωση του όγκου των φυτοφαρμάκων ε, θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση εναλλακτικών λύσεων γιατί υπάρχουν κάποιες ε, ουσίες που δεν θεωρούνται φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά χρησιμοποιούνται για τη φυτοπροστασία, ενώ η χρήση τους εξαρτάται, από το κανονισμό 1107 το 79, που ίσως ε, αποτελέσουν τελικά εναλλακτική λύση αν ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Επίσης υπάρχουν πολλά προϊόντα που άπτονται του βιοελέγχου. Ενδιαφέρουσες λοιπόν όλες αυτές οι διαδικασίες. Έχουμε και μη χημικές μεθόδους ε, για την πρόληψη πολύ πιο φιλικές ε, στην υγεία και το περιβάλλον από τα φυτοφάρμακα. Οπότε, ε, καλό θα ήταν να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των διαφόρων μεθόδων ε, και των χημικών μεθόδων. Για παράδειγμα, αμυψισπορά που ανέφερε ο κύριος Χόσλινγκ, αλλά και ε, αξιολόγηση των μηχανικών μεθόδων. Επίσης, θα πρέπει να λεφθούν υπόψη οι συγκριτικέ αξιολογήσεις κατά τη θέση εμπορία των σκευασμάτων, όπως πρότειναν η κυρία Αντριό και Νταντά. Οι γεωργοί παραπονιούνται για την έλλειψη εναρμόνιση σε ό,τι αφορά τη θέση σε εμπορία των προϊόντων, γιατί μερικά προϊόντα φυτοπροστασία κυκλοφορούν σε ορισμένε χώρε και όχι σε άλλε, δημιουργώντα τρέβλου ανταγωνισμού μεταξύ των ε, Ευρωπαίων γεωργών. Και μάλιστα υπάρχει και μερικέ φορέ λαθρεμπόριο διασυνοριακό τέτοιων προϊόντων. Κυρία Χόιμπουχ. Ε, ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ πρέπει να πω ότι εξεπλάγει και κατεπλάγει από τα όσα είπε ο κύριος ε, Άνιου το ότι μπορεί να καταπιεί ένα ζενιοκτόνο σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να τον οδηγήσει σε θάνατο είναι απαράδεκτη δήλωση βεβαίως έχουμε πολύ ακραίες δηλώσεις εδώ εδώ βλέπουμε στην γνωμοδότηση λοιπόν ότι δεν θα πρέπει η αδειοδότηση να στηρίζεται σε φοβικές αντιδράσεις αλλά στην επιστήμη. Όταν όμως έχουμε τον πληθυσμό ο οποίος ανησυχεί γενικότερα και να το ε, ε, ε, εξαντλούμε αυτό σε μια δήλωση ότι πρόκειται για φοβικές αντιδράσεις γιατί βεβαίως και αυτές οι επιφυλάξει των πολιτών στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και πρέπει να τις εισακούσουμε αυτές τις ανησυχίες. Ε, διαφορετικά νομίζω ότι είναι κατανοητό το γιατί πώς τόσοι πολίτες εγκαταλείπουν, την πολιτική, εγκαταλείπουν το ενδιαφέρον τους για την πολιτική. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επιστημονικά δεδομένα και διαφάνεια σε σχέση με το πώς προκύπτουν οι επιστημονικές αυτές μελέτες κατά τρόπο ανεξάρτητο από επιστήμονες ανεξάρτητος και και με τρόπο επαληθεύσιμο. Ε, και αυτό, όχι και το είπε πολύ καλά ο κύριος Χόισλινγκ, διότι έχουμε ε, κάποια επιφυλεκτικότητα, αλλά γιατί υπάρχουν όντως διαφορετικές βάσεις για μια επιστημονική έρευνα και πρέπει να επικρατήσει η αρχή της πρόληψης και της σύνεσης. Ας μην αφήσουμε λοιπόν να χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Εμπιστοσύνη που χρειάζεται και ο Γιώργος και η γεωργική πολιτική. Άννα διαμορφώνεται η γεωργική παραγωγή κατά τρόπον ώστε ο πολίτης πλέον να μην έχει εμπιστοσύνη, τότε η ζημιά φτάνει μέχρι και τον γεωργό. Ε, ο πολίτης ο οποίος καθημερινά αγοράζει το τροφιμά του για τη διατροφή του πρέπει να αισθάνεται εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο τι χρειαζόμαστε για τη γεωργία σήμερα δηλαδή όλο και πιο εξορθολογισμένη παραγωγή, μέγιστη δυνατή παραγωγή και συγκομιδή, τι είδους γεωργικά συστήματα χρειάζονται πιο μέσων για να λειτουργούν χωρίς όμως ανεβιώσιμα κοινωνικά. Αυτό δεν μας οδηγεί πουθενά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Οι παρατηρήσεις σας επί της γνωμοδότησης ΓΙΑΡ φαντάζομαι καταγράφονται και θα διαβιβαστούν ε, στον αρμόδιο από τον κύριο Ντές, ο οποίος έχει και το λόγο αν θέλει να σχολιάσει μετά από τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους ε, που συνέβαλαν στη συζήτηση, τους κοιόδης ηγητές και συγητρίες. Βεβαίως θα διαβιβάσω όλα τα στοιχεία στον Πετριάρα, άλλωστε και οι συνεργάτες του είναι εδώ και τα έχει καταγράψει όλα. Αλλά επιτρέψτε να δώσω κάποιες απαντήσεις στις παρατηρήσεις. Ε, μόλις έλαβα στοιχεία από τη Γερμανία, Το 2016 χρησιμοποιήθηκαν 3.780 τόνοι γλυφοσάτη στην Γερμανία, ε, κατά το ίμιση στην ε, Γεωργία και κατά το ίμιση από ό,τι λέγεται από τους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Είχαμε πριν από χρόνια όμως 60% περισσότερο, μεγαλύτερο όγκο χρησιμοποιούμενης από τη γεωργία γλυφοζάτης. Επομένω, πιστεύω στο μέλλον και για λόγους τεχνικούς ακόμη θα έχουμε ε, ανάγκη για λιγότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Προχωρεί μια τεχνολογική επανάσταση στα θέματα αυτά και ήμουν στο Βερολίνο στην πράσινη λεγόμενη εβδομάδα όπου με εντυπωσίασαν τα πόσα μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία για το μέλλον της γεωργίας με ε, αποτελεσματικότητα το 80% μεγαλύτερη από δραστικές ουσίες σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα. και πιστεύω ότι ήμασταν πολύ από τη Γεωργική Επιτροπή, αλλά και ο κύριος Δεκάστρο στο Birmingham, όπου συζητήσαμε τα θέματα που φορούσαν την ε, πατάτα και τη δυνατότητα για στοχευμένη, με πολύ περιορισμένη χρήση ε, δραστικών ουσιών, μέχρι, και 10, μέχρι στο 10% δηλαδή, δραστική ουσία μπορούσε να αντιμετωπίσει το ε, πρόβλημα που μπορούσε να παρουσιάζει το προϊόν. Ε, η τεχνολογία λοιπόν σύγχρονη έχει πολλά να μας προσφέρει. Για την κυρία Αγγιλέρα τώρα θα ήθελα να πω, αλλά και ο κύριος Ντόμπτο. Είπαν ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μια ευρωπαϊκή αρχή αδειοδότησης. Δεν είναι δυνατόν από 28 κράτη-μέλη ε, το καθένα να κάνει τη δουλειά στη γωνιά του και εν τέλει να μην υπάρχει ένα ε, ενιαίο αποτέλεσμα. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καλύτερα αποτελέσματα Ούτε μπορεί βέβαια να γίνεται έρευνα σε 28 διαφορετικά κράτη-μέλη χωριστά, γιατί αυτό σημαίνει και πολύ ε, περί κόστος και δαπάνες για την έρευνα. Έγινε λόγος, ε, υποστήριζω προσωπικώς όλους τους συναδέλφους ε, που έθιξαν το ζήτημα αυτό της ανεξάρτητης έρευνας, που οπωσδήποτε θα κερδίσει και πιστωρή υποδοχή από τους πολίτες. Έχω μάλιστα τα τελευταία στοιχεία για τα ζεζανιοκτώνα και τις πολυματικές ουσίες τους ε, στα φύτα για το 2016 συγκεκριμένα 19.899 δείγματα που εξέτασαν στα εργαστήριά τους ε, τα κράτη καταγράφουν με 5,8 εκατομμύρια αναλύσεις, 1,7% των δειγμάτων που εξετάστηκαν, δειγμάτων τροφίμων, καταγράφουν χαμηλή ε, χαμηλό ποσοστό υπέρβασης των ε, οριακών τιμών. Ενώ σε εισαγωγέ από τρίτα κράτη, όχι Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αλλά τρίτα κράτη, έχουμε 6,3% αντίστοιχε τιμέ υπέρβασης εισαγωγές από την Ταϊλάνδη, τη Σριλάνκα νεροσπανακιού μας δίνουν ε, υπέρβαση έως και 56%. Ε, έτσι λοιπόν έχουμε να σημειώσουμε ότι στα κράτη-μέλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Οι δε υπερβάσεις με ύψιστη στον Αρακά, στα άγρια μανιτάρια, είναι 2,4% μόνο. Και ας δούμε ποια είναι τα ζυζανιοκτώνα ή τα αυτοπροστατευτικά χαλκός 2,6%. Τάτσετη Μιμπρίδιου με 2,9%. Εδώ έχουμε να κάνουμε με, τα, με ουσίες οι οποίες είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ως φυτοπροστατευτικές και για τη γλυφοζάτη Είχαμε 4.048 δείγματα, 0,3% πάντα στο 2016 σημειώνουν ε, υπέρβαση των οριακών τιμών ε, στο μέλι και σε, άλλες σε άλλα προϊόντα, πάρα πολύ χαμηλά δηλαδή ποσοστά υπέρβασης. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει τι είδους ε, συζήτηση και πού εστιάζουν ορισμένοι τη συζήτηση. Επίσης, είχαμε κατά το μεσαίωνα τεράστια προβλήματα ε, και μάλιστα στη Γαλλία πριν από την Γαλλική Επανάσταση 20.000 νεκρούς λόγω της ε, ε, επιμόλυνσης με μύκητες που είχε προξενήσει η, η υγρασία. Μέχρι το 1900 δεν είχαμε, μέχρι το 19ο αιώνα δεν είχαμε φυτοπροστευτικά προϊόντα, μέγιστο, μέγιστο προσδόκιμο ζωής 39 χρόνια ζωής ε, στη Γερμανία, ενώ τώρα έχουμε φτάσει στα 80, κάθε χρόνο ανεβαίνει αυτό το προσδόκιμο κατά 3-4 μήνες στη Γερμανία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι η συζήτηση ε, η οποία έχει οδηγήσει σε μια δαιμονοποίηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι τελείως εσφαλμένη. Βεβαίω πρέπει να γίνονται ανεξάρτητε έρευνε από ανεξάρτητου επιστήμονε, Αλλά όχι από αυτού οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για την ε, χρήση και τα αποτελέσματα των φυτοπροστατευτικών. Και όπως είπα, η νέα τεχνολογία θα μας εξασφαλίσει ακόμα πιο θετικές συνθήκες και αποτελέσματα. Προς το παρόν όμως τα φυτοπροστατευτικά τα χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο προστασίας των φυτών μας, όχι με υπερβολές, με τα σωστά μέσα και για τον κύριο Ανιού θα ήθελα να αναφέρω το... να απαντήσω στο ερώτημά του για, τις 160... για το 140 ημέρες ότι ναι είναι μια προθεσμία που θα πρέπει να τηρείται μέρος του κυρίου Κύριε Ευρωβουλευτά δεν ξέρω αν είχατε την έγκριση του κυρίου Γιάρ για να απαντήσετε τόσο διεξοδικά σε όλες τις ε, παρατηρήσεις γιατί πραγματικά απαντήσατε σαν να ήσταν εισηγητής. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώ ε, ολοκληρώσαμε αισίω τη συζήτηση. Μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να υποβάλλετε τις τροπολογίε σας και ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό. Αύριο σε 9 θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορίες. Παρακαλώ μην ξεχάσετε τι κάρτε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ. Σήμερα ήταν πολύ χαλαρό το απόγευμά μας και έτσι είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου και δεν χρειάστηκε να διακόψουμε τους συναδέλφους. Καλό σας ε, απόγευμα βράδυ. Τέλος της συνεδρίασης.